Ε, του, κανονισμού για τα ευρωπαϊκά δεδομένα, ούτω ώστε στο έδαφο τη Ευρωπαϊκή Ένωση να εφαρμόζεται το ευρωπαϊκό δίκαιο. Ευχαριστούμε θερμά, κυρία Επίτροπε. Ε, ε, ε τελειώσαμε, ε, ήλπιζα να τελειώσουμε πριν από τις 12, τελειώσαμε έγκαιρα, ευχαριστώ τους πάντες, ε, τους συνεργάτες μας και τους διερμηνείς. Ε, ολοκληρώσαμε την διαδικασία και ε, θα συνεχίσουμε από ε, τις 9 μέχρι τις 12, 5 16 Φεβρουαρίου. Είναι στην διάθεσή μας, θα είναι στη διάθεσή μας τα πρακτικά. Ολοκληρώσαμε τη συνεδρίαση. Καλό σας βράδυ.